Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. uh, a Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 14ης Οκτωβρίου. Το πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης ε, είναι φυσικά η έγκρισή της. Οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, την εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, μία μόνο ανακοίνωση. Η, αποφα... η αποφάση των συντονιστών της 30 Σεπτεμβρίου 2019 θα υπάρχουν στα πρακτικά, στα... στο φάκελο με τα έγγραφα της συνεδρίασης. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσει και για αυτές θα θεωρηθούν συγκεκριμένε. Επίση, Επίσης, έγκριση των πρακτικών της 24 Σεπτεμβρίου και πάλι αν δεν υποβληθούν αισθάσει θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Ωραία. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε πρώτα τον προϋπολογισμό του 2020. Καταρχήν να δοκιμάσουμε τις ε, συσκευέ τα μηχανήματα της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εντάξει, λειτουργεί το σύστημα. Ήταν δοκιμαστική η ψηφοφορία, είπαμε. Περνάμε τώρα στο κατάλογο ψηφοφορίας. Πρώτα θα ψηφίσουμε διανατάσταση της χειρός. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. 13. 1-3. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 13. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Ποιο... Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Κανείς. Εγκρίνεται. Αποχές. Αποχές λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Τροπολογία 55. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 10 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 75. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μα, κατά. Πρώτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Κανένα πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λάθος με ακούλπα. Συγγνώμη. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια δυστυχώς. Λυπούμε, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε ή 82 εγκρίνεται. 83 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα μόνο της τροπολογίας 84. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote open. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. This is withdrawn. Amendment 89. Τροπολογία 89. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Everybody voted. Vote closed.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 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 106. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 και 113 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. 112 και 113 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 17 της ΑΦΕΤ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφέτη 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115. Λαγός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αύκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 129 Everybody voted Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132. 132. Έχει αποσυρθεί. 133 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελογίας παράγραφη παριθμών 1 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Παριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περιθμόν 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια για την κυρία Χόλμαγερ. Και την κυρία Γκουαρντιθάβαλτση. καταληκτικές παρατηρήσεις, οι, οι διάλογοι ε, έχουν προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου. Η συζήτηση και η έγκριση στην Ολομέλεια για τη θέση του Κοινοβουλίου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, 23 Οκτωβρίου. Και η πρώτη συνεδρία συνάντηση συνδιαλλαγή έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου στο Κοινοβούλιο στις 5 το απόγευμα. Και τώρα. Πέντε. Μόλις λάβαμε το σχέδιο εγγονισμού του Συμβουλίου, που αφορά το σημείο 5, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σήμερα και διαβιβάστηκε στους συναδέλφους. Έχουμε πάρα πολλές ευθρέουσες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε σας προτείνω να ψηφίσουμε ούτω ώστε να ψηφίσει η Ολομέλεια για όλα τα κατεπηγόντα μέτρα σε σχέση με το Brexit στην Ολομέλη την άλλη εβδομάδα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Έξι. Τμήμα 3. Μεταφορές. Προτείνω στον κύριο Χάουαρθ να μας εξηγήσει ένα-ένα τα τρία αυτά σημεία. Πρώτα το 10-16. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε τρεις ε, αιτήσεις για αυτή την μεταφορά, 16, 17 και 18. Το DEC. Το 16 είναι η πιο σημαντική ε, συνολική μεταφορά. Γίνεται συνήθως τέτοια εποχή. Είναι δημιουργικά ουδέτερες αυτές οι μεταφορές, ούτε αύξηση, ούτε μείωση. Έχουμε. Εδώ είπαμε ότι από το 22-26 θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά και αφορά κάποιες πιστώσεις πληρωμών. Γαλιλαίο, έγνος, έρασμος, συν και η εκτέλεση προχώρησε πιο γρήγορα από όσο προβλεπόταν. Οπότε αυτά αντισταθμίζονται από κάποιες μειώσεις της υποχρεώσεις από πέντε κονδύλια και που είχαμε πιο αργή εκτέλεση και καλύπτονται ένα σώρο κονδύλια και συγκεκριμένα το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το HCP και κάποια κομμάτια του Horizon 2020. Αυτά είναι στην πρώτη σελίδα του σχετικού εγγράφου. Και εκεί αναφέρονται συνοπτικά αυτές οι μεταφορές, στο σύνολο είναι ένα δις 77.588.000. πολλά χρήματα, αλλά αυτό είναι μια μικρή απόκληση από ένα 0,7% από τι εγκριθήσει πληρωμές για το 19. Το σύνολο τη μεταφορά για το 19 είναι περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό το πολιτεύει δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί όπω όλοι ξέρετε τώρα, πλησιάζουμε το τέλο αυτού του πολιτικού πλαισίου και επομένω έχουμε αυτήν την αύξηση σε δύο τομείς όμως θα πρέπει να μας κάνει ε, σχετικά σχόλια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξηγήσει λίγο περισσότερο που λένε τα έγραφα. πρωτα Πρώτα-πρώτα το γενικότερο θέμα. πόσο δηλαδή αυτέ οι μεταφορέ, αυτέ οι πληρωμέ έχουν κάποιε συνέπειε για το 2020. Τέλο του τωρινού πολιτικού πλαισίου και δεύτερον, όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Άμυνα, εδώ είναι ένα ε, τομής που έγινε το θαύμα, βρέθηκαν οι αρχές και έτσι το πρόγραμμα μπόρεσε να ξεκινήσει αρχές του 19. Επίσης, σύμφωνα με τη σελίδα 4 της έκθεσης, δεν είχαμε κάποιο είδους συμφωνίες και το πρόγραμμα αυτό για την άμυνα πήγε το 2020, να μας το εξηγήσει η Κομισιόν. Και, Πρόεδρε, προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση αυτής της ε, συνολικής μεταφοράς. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Άλλος από τους συναδέλφους. Then I think we can proceed. Δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση. Κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you to the rapporteur for the uh, support ευχαριστήσω τον εισηγητή που εκφράσει την υποστήριξή του mm. στη σημαντική αυτή μεταφορά. Δύο ερωτήσεις νομίζω είχατε, κύριε εισηγητά. Η πρώτη είναι η γενική ερώτηση, δηλαδή ποιος είναι ο αντίκτυπος της μεταφοράς αυτής στο επίπεδο των ε, ε, πιστώσεων πληρωμών για το 2020. Γενικά, η έγκριση της μεταφοράς αυτής ε, δεν ε, αναμένεται να επηρεάσει το συνολικό ε, επίπεδο των πληρωμών για το 2020, διότι είναι ουδέτερη για το 2019 και θα είναι ουδέτερη και το 2020. Χάρη σε αυτήν την μεταφορά θα έχουμε και καλύτερη υλοποίηση εντός του 2019, δεν θα έχουμε δηλαδή υποεκμετάλλευση στην άμεση διοίκηση, όπως θα συνέβαινε σε διαφορετική περίπτωση και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταφορά πιστώσεων προς διαχείριση. Με αυτή λοιπόν τη γενική μεταφορά θα μεταφέρουμε κάτι περισσότερο ε, για το 2020. Αλλά γενικώς ουδέτερη είναι αυτή η μεταφορά. Άρα δεν χρειάζεται άμεσα να αναθεωρηθούν ε, τα επίπεδα πληρωμών όπως προτείνονται αυτά από την Κομισιόν στο σχέδιο προϋπολογισμού που έχει καταθέσει. Σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο ερώτημα που κάνατε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της αμυντικής βιομηχανίας ε, είναι διετούς διάρκεια. Συγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου του τρέχοντος. Έχουν ε, προκηρυχθεί έκτοτε εννέα διαγωνισμοί και σε ό,τι αφορά ε, για αυτές τις νέα προτάσεις ε, το τέλος της προθεσμίας ε, ήταν ο Αύγουστος. Είναι πολύ πλοκό όμως αυτό το πρόγραμμα, οπότε οι υποψήφοι με την υποστήριξη των μελών ζήτησαν παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για αυτούς τους διαγωνισμούς. Η Κομισιόν λοιπόν δεν έχει μπορέσει μέχρι τώρα να αξιολογήσει, να υπογράψει συμβάσει και να κάνει τις πληρωμές πριν τα τέλη του τρέχοντο. Δεν θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο, άρα θέλουμε προχρηματοδότηση, προκαταβολή. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 προβλέπεται αυτό. Για να αποφύγουμε όμως να έχουμε τα ίδια και το 2020, προτιθέμεθα τις επόμενες προκηρύξεις ε, να τις ε, δρομολογήσουμε ήδη από το Γενάρη του 2020. Άρα πρώτες πληρωμές για τους διαγωνισμούς 2020 θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα λάβουν χώρα στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 και ελπίζω να απαντώ στο ερώτημά σας. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει σχόλια ή να συμπληρώσει κάτι. Κύριε Πρόεδρε, κύριο Χόρθ, να εγκρίνουμε, θα έλεγα τότε, αυτή τη μεταφορά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα χωριστά της ΔΕΚ 17, 18, 19, λέει ο πρόεδρος. Oh, Α, με συγχωρείτε, δεν έχετε παρουσιάσει τις άλλες δύο μεταφορές. Ναι, όπως θέλετε, να ψηφίσουμε την πρώτη, να ψηφίσουμε μαζί. Ωραία, ας ψηφίσουμε τώρα την πρώτη, λέει ο πρόεδρος. Άρχεται ονομαστική ψηφοφορία για τον ΔΕΚ 16. Ποιος είναι υπέρ. Ναι, είναι Δευτέρα, τι να κάνουμε. Τέλο πάντων, πέρα ψηφοφορία. Να ξαναρχίσουμε, γιατί σας μπέρδεψα και τα μπέρδεψα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Λυπούμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Χάουερ. Για το 17. Of the European Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονία. 50,7 εκατομμύρια ευρώ σε, δεσμό, ε, σε ανάληψη υποχρεώσεων για να μπορέσει να έχουμε δράσει στον τομέα τη διαχείριση στο Μαρόκο και να ενισχύσουμε την προστασία μεταναστών προσφύγων κτλ. στη Λιβύη. Έξι κονδύλια του προβλησμού θα χρησιμοποιηθούν, ιδίω μάκρο χρηματοδοτική βοήθεια, ενίσχυση ε, και ε, αποστολές παρατηρητών σε εκλογές. Σε ό,τι αφορά το είδο των δραστηριοτήτων που προτείνονται για το μέσο για το Νέα Σιλιβή και Μαρόκο, θα θέλαμε κάποιε παραπάνω πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Και για την ετοιμότητα αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε τρίτε χώρε 23 03 αν δεν ε, είναι ποιοτικέ οι προτάσεις, επαρκείς προτάσεις, ε, πώς θα βελτιωθεί αυτό η κατάσταση των προτάσεων δεν δηλαδή είναι ποιοτικέ ε, και έτσι θα έχουμε καλύτερη διαχείριση στο Θα περιμένω να απαντήσει η Κομισιόν και μετά θα σας πω αν θεωρώ ότι πρέπει να εγκρίνουμε όχι τη μεταφορά η Κομισιόν. Uh, thank you, and thank you to the for... Ευχαριστώ πολύ σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε που θα ενισχυθούν με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονία, Τα 5,7 εκατομμύρια που θέλουμε παραπάνω στις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων θα συνιστούν μια συμβολή του ίδιου ποσού στο βορειοαφρικανικό σκέλος ε, του καταπιστεύματος της Αφρικής για να κλείσει ένα κενό, μια τρύπα στη χρηματοδότηση που εντοπίσαμε σε ό,τι αφορά τις ε, δραστηριότητες που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν εντός του 19. Συγκεκριμένα λοιπόν, με αυτά τα χρήματα θα έχουμε, όπω είπα, χρήση του καταπιστέματος της Βορειοαφρικής για το Μαρόκο δραστηριότητες διαχείρισης συνόρων. Δεύτερον, στη Λιβύη ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων ε, που είναι στη χώρα αυτή εγκλωβισμένη και θέλουμε να βρούμε επίσης εναλλακτικέ λύσεις αντί της παράνομης ε, κράτησης ή της προσωρινής κράτησης. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τις προσπάθειες σταθεροποίησης δίνοντας μεγαλύτερη υποστήριξη σε δήμους, κοινότητες και ευάλωτους πληθυσμούς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα κάποιος το λόγο από την Επιτροπή μας. Αν όχι, να ξεκινήσει η ψηφοφορία, παρακαλώ. Vote closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Χάουερτ, για τον ΤΕΚ 19. Finally, Οπότε, στο 19 έχουμε έτοιμα μεταφορών 530.000 ε, ε, μεταφορά ευρώ σε επιστώσεις αναλήψης υποχρεώσεων και επιστώσεις πληρωμών από την, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Χημικών Ουσιών, το ΕΧΑ. Και επίσης θα έχουμε ανάληψη υποχρεώσεων από τις μεταφορές και μεταφορά από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, γιατί χρειάζονται να αντισταθμιστούν οι αυξήσει του κόστου προσωπικού εν μέρη σε κακό υπολογισμό του κόστους μισθών και σε προβλέψεις για τη μελλοντική στελέχωση. Πάντως δεν έχω συμπληρωματικές ερωτήσεις για τη σχετική μεταφορά. Θα ήθελα απλώς να σας συστήσω την έγκρισή της. Θέλει κανείς το λόγο για να σχολιάσει την πρόταση του εισηγητού. Όχι, οπότε ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή η μεταφορά. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Μεταφορές του 2019. Λοιπά τμήματα. Ο, ο συνάδελφος Φερνάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ μία μεταφορά για την ΑΕΔ και τέσσερις για το ελεκτικό συνέδριο. Θα σας τις παρουσιάσω από κοινού αυτές τις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι μεταφορές οφείλονται στην αύξηση των αρμοδιοτήτων ε, της ΑΕΔ. Και αυτή η πρόταση μεταφοράς από ανάληψη υποχρεώσεων αφορά 2,3 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ε, στελέχωσης, ε, των μέτρων για τα κτίρια, οπότε αφορά στήλες και το μη σχετικά ζητήματα, ε, τα συνέδρια της διασκέψης και τις υπηρεσίες πολυγλωσσίας. Αυτές οι μεταφορές οφείλονται από οικονομίες, οφείλονται σε οικονομίες που έγιναν σε άλλες δημοσιονομικές γραμμές. Σε ό,τι αφορά το ελεκτικό συνέδριο τώρα και τη μεταφορά 13, 6.000 ευρώ για μετακομίσεις και συναφή κόστος και 22 επίσης ευρώ για σύστημα συνδιαχείρισης και διενέργειας ελέγχου. Και το ποσό αυτό προέκυψε από το άρθρο 214 που αφορά το τεχνικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Άλλη μεταφορά για το ελεκτικό συνέδριο. Είναι υπαριθμό 14 ύψους 4.000 ευρώ. Για την ενίσχυση του συστήματος συνδιαχείρισης και ελέγχου και για την ε, για το πρόγραμμα ε, που εμπνέει περισσότερη βιωσιμότητα. Και τώρα ε, θα προκύψει από το 29 ε, λοιπές δαπάνες. Άλλη μεταφορά είναι η μεταφορά υπέρθυμα 15 από το στοιχείο 2720 με τίτλο «Δαπάνες ε, για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση και τα αρχεία. 10.000 ευρώ είναι το ύψος της μεταφοράς αυτής. Και επιτεύχθη χάρη σε οικονομίες από το 2070 από την γραμμή 2073. Και τέλος, η παριθμό 16 η ε, μεταφορά είναι ύψος 30.000 ευρώ για έπιπλα, επίπλωση και προήλθε από εξοικονόμηση ε, στο 2300 με τίτλο «Εξοπλισμός γραφείου, και αναλώσιμα». Εγώ προτείνω να υπερψηφίσουμε αυτές τις πέντε μεταφορές, μία για την ΕΕΔ και τέσσερις για το ελεκτικό συνέδριο. Συνολικά δηλαδή πέντε μεταφορές, τις οποίες αισθήνω να υπερψηφίσουμε. Μάλιστα. Θέλει κανείς το λόγο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνουμε τις μεταφορές και τις πέντε που μας, σύστησε, μας παρουσίασε και μας σύστησε να υπερψηφίσουμε ο κύριος Φερνάντες. Και συγχαρητήρια κύριε Φερνάντες. Σημείο 8. Κτηριακή πολιτική. Δεν έχουμε στο πρόγραμμα θέματα σε σχέση με κτίρια, οπότε ολοκληρώνουμε τις ψηφοφορίες μας για σήμερα. Συνεχίζουμε στο σημείο 9 που αφορά και πάλι κτηριακή πολιτική, αλλά ούτε και εδώ έχουμε φαγγέλους για θέματα κτίριων. Σημείο 10. Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπια. Αφορά μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορο... Ε, με προϋπολογισμό συγγνώμη, στην αρμόδια κατουσία επιτροπή που είναι η Επιτροπή Αλίας και που πρόκειται να εκπονήσει μια σύσταση για συγκατάθεση σε ό,τι αφορά το κανονισμό του Συμβουλίου βάσει νομοθετικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την διμερή, τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, εν προκειμένου ε, της Γκάμπια, στα θέματα της βιώσιμης αλίας και μάλιστα περιλαμβάνεται και ένα πρωτόκολλο που καλύπτει τις οικονομικέ ε, οικονομικές συνεισφορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σαστέλ που θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση αυτής της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Γκάμπια. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Κύριε Σαστέλ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε εμείς θα, θα, δώσουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ελίε για την ανανέωση της Συμφωνίας Σύμπραξης βιώσιμη Ελίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γκάμπια και γνωμοδότηση για το πρωτόκολλο εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τι διαπραγματεύσει για τον προσδιορισμό ε, των δυνατοτήτων αλληλεία Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικονομικό αντάλλαγμα για την αλληλεία στα χωρικά ύδατα τη Γκάμπια. Παρακαλώ, λίγο σεβασμό προ τον συνάδελφο, τον κύριο Σαστέλ. Λίγο σεβασμό, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, λοιπόν. Στις 19 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και μονογράφηκε η ανανέωση της συμφωνίας και το νέο πρωτόκολλο. Και μάλιστα ε, η ανανέωση γίνεται σιωπηρά και το νέο πρωτόκολλο καλύπτει μια εξαετία από το 2019 στο 2024 και εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής. Στόχος της νέας συμφωνίας είναι η επικαιροποίηση του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ και της εξωτερικής διάστασής της, προκειμένου να σφυριλατηθεί στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γκάμπια στα θέματα τη Αλία. Το πρωτόκολλο επίση δίνει ένα νέο δυναμισμό στη συνεργασία με τη χώρα αυτή και συσφίγγει τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Γκάμπια προκειμένου να εφαρμοστεί μια βιώσιμη ελεία και μια υπεύθυνη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ελευτικών πόρων στα χωρικά ύδατα της Γκάμπια. Και φυσικά η τεκμηρίωση προκύπτει από επιστημονικά πορίσματα και πρόκειται για μια αμοιβαίως εποφίλη προσέγγιση γιατί και τα, δύο και τα μέρη συμφώνησαν για τους όρους που διέπουν την αλία από ευρωπαϊκά σκάφη στα χωρικά ύδατα τη και καθορίζεται και η κοινοτική συνεισφορά προκειμένου να ενισχυθεί βιώσιμη αλληλεία Πρόκειται για 550.000 ευρώ ετησίω, ε, δηλαδή 3,3 εκατομμύρια για το σύνολο τη εξαετία. και ε, κάθε χρόνο ε, δαπανώνται 275.000 ευρώ για την πρόσβαση στους ελευτικούς πόρους στα ελευτικά πεδία της ε, Γκάμπια, δηλαδή 3.300 τόνοι ετησίως και μάλιστα υπό επιφύλαξη του κόστους πρόσβασης που είναι 315.000 ευρώ το χρόνο και το αναλαμβάνουν οι εφοπλιστές και επίσης στήριξη της τομεακής πολιτικής της Γκάμπια, πάλι το ύψος είναι 275.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Γκάμπιας να εφαρμόσει μια βιώσιμη πολιτική αλίας με την τομεακή αυτή στήριξη και λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους. Η νέα συμφωνία λαμβάνει υπόψη και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως το άρθρο 9 της συμφωνίας Κοτονού με βάση λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια, θα ήθελα να σας προτείνω να υπερψηφίσουμε τη γνωμοδότηση, συστήνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου και για τη σύναψη Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας, καθώς και το νέο πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Θέλει λόγο από Τότε απλώ προσθέτω ότι σας επισύρω την προσοχή ότι σε μια τέτοια συμφωνία συνειδητική χωρίς ψήφισμα ε, ε, νομοθετικό από την κύριο Σωματεπιτροπή μόνο έγκριση ή απόρριψη ε, προβλέπονται. επομένω δεν προβλέπονται τροπολογίες. Θα γίνει η ψηφοφορία στις 6 Νοεμβρίου. Οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο 11 κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχει το λόγο εισηγητής ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ή Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα ταμείο που στηρίζει τους ε, ε, εργαζόμενους που έχασαν την θέση τους λόγω της παγκοσμιοποίησης και έχουν πληγεί από αυτή. Και Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό ταμείο. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα άλλα ταμεία. Ούτε έχει στόχο το ταμείο αυτό να υποκαταστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι ε, επικουρικό, συμπληρωματικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στο Carrefour, στο σούπερ Carrefour του Βελγίου. 1.632.028 ε, ευρώ είναι το ποσό που προτείνεται να ενεργοποιηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης και θα βοηθήσουμε έτσι 1019 εργαζομένους στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ Carrefour, είτε μέσω δράσεων για την ε, ε, επιστροφή στην αγορά εργασίας ή ε, διάφορες δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και επίσης προβλέπει υποστήριξη για αυτοαπασχόληση, για τη δημιουργία νεοφιών επιχειρήσεων. Πολλές θέσεις ε, εργασίας χάθηκαν στα σούπερ μάρκετ Carrefour. Ε, λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι έκλεισαν πολλά σούπερ μάρκετ και περιορίστηκε δραστικά ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο αυτό. έχουμε ε, το 80% των εργαζομένων αυτών να είναι 55 έως 64 ετών. Επίσης ε, προέρχονται από τη Βαλονία που έχει υψηλό ποσοστό ανεργία περίπου 12,6% πολύ πάνω από το κοινοτικό μεσόρο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το σχετικό κονδύλιο από το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχε περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το ποσό που σας ανέφερα για τη στήριξη αυτών των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Carrefour. Ο πρόεδρος, κύριος Ζάκοφ. Γενικά είναι μεγάλη η πρόκληση, αλλά θα πρέπει να μπούμε στι λεπτομέρειε. Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να καλύψουμε πολλές κρίσεις όσον την απασχόληση λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ε, πρόοδου της τεχνολογίας, οπότε έχουμε κάποιες τροπολογίες, ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να είναι πιο στεγανό το έγγραφο. Κύριε Σώστελ, ευχαριστώ. Φυσικά και συμφωνώ με τον εισηγητή μας. Νομίζω ότι τα εξήγησε σαφώς αυτό το οποίο εδώ ζητείται από το Βέλγιο κατόπιν τη ε, απόλυση πάνω από χιλίων εργαζομένων από το Καρφούρ. Αυτό πρόκειψε σε μία περιφέρεια. Έχουμε 400 που απελευθερία, αλλά έχουμε και 300 νέους κάτω από το, τα 25 που δεν έχουν ε, κάποια κατάρτιση, δεν σπουδάζουν, οπότε τώρα μπορούν να έχουν κάποιες προσωπημένες υπηρεσίες ε, προσανατολισμού επαγγελματικού, οπότε έτσι θα έχουμε 2.300 ε, ευρώ για αυτούς τους 530 εργαζομένους, όπως είπε και η Μαρία Τάση είναι επίτροπο για την απασχόληση. Είναι πολύ σημαντική η κοινοτική ελεγγύη για να καλυφθούν οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι. Όντω, όπω είπε ο συγητή, στη Βαλονία έχουμε ιδιαίτερα υψηλή, ιδιαίτερα αυξημένη πάνω το μέσο όρο ε, ανεργία και το 2018 στους ανέργους είχαμε 22,5% ανεργία. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ακόμα ένας λόγος για να ληφθεί υπόψη αυτό το αίτημα γιατί ε, αφορά αυτούς τους 330 νέους οι οποίοι έτσι θα έχουν ε, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικό ανατολισμό ε, και έτσι θα μπορούσαν να ψάξουν για δουλειά. Οπότε και εγώ συμφωνώ με τα όσα συνεπέραν ο εισηγητής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει άλλο συνάδελφο το λόγο. Αν όχι, τον, θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να πανεύω εκτός από το να ευχαριστήσω τους βουλευτές και τον εισηγητή και να διευκρινίσω αυτό το μυστηριώδες 18 και ο κύριο Χάουαθ ε, αναρωτιόταν ακριβώς ε, τι, τι μεταφορά πίστοσης είναι αυτή ε, για το Καρφούρι. Κύριε Φεράντες, θέλετε κάτι να παρατηρήσετε. Ευχαριστώ Όσο έλαβαν το λόγο. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε διάφορες κινητοποίησεις του Ταμείου προς την ίδια κατεύθυνση. Η δε προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 22 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η ψηφοφορία προβλέπεται να γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ και προχωρούμε στο σημείο παρασμό 12. Mrs. Holmeyer has disappeared. Έφυγε όμως η κυρία Χολμαϊρ. Α, θα εμφανιστεί. Θα επανεμφανιστεί, οπότε ο λιγόλεπτη διακοπή. Uh, Είμαστε στο σημείο 12 της ημερησίας διατάξεως όσον αφορά το Ταμείο Ελληνικής. Και ε, ευχαριστώ σας δίνω τον ε, λόγο κυρία Χολμαϊρ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την κινητοποίηση. Το Καρφούρ. Α, λάθος. Για να αλλάξω θέμα κινητοποιεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Βέλγιο, το Καρφούρ, όχι. Συγγνώμη, έχω τελείως λάθος χαρτιά μπροστά μου. Γιατί έβλεπα Ταμείο Αλληλεγγύης, μα Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, ναι, εγώ θέλω να πω για την πρόταση της Κομισιόν για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να είναι ευέλικτη και να χρησιμοποιείται το Ταμείο αυτό όταν χρειάζεται. 50 εκατομμύρια είναι το ανώτατο ποσό για τις προκαταβολές, 10% δηλαδή. Τώρα, ε, κατά πόσον βοηθά ε, να έχουμε λίγο παραπάνω επίπεδο προκαταβολές είναι υποσυζήτηση. Ε, το Ταμείο Αλληλεγγύης πάντως πολλές φορές πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα οι πολύπλοκες διαδικασίες για την υποβολή αιτημάτων και αυτό νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ναι. 10% λοιπόν είναι το ανώτατο ποσό. Ούτω ή άλλω ο προπολογισμό είναι 500 εκατομμύρια και το μέγιστο αυτό ποσό δεν πρέπει να ε, ξεπεραστεί. Υπάρχουν 15 αιτήματα μέχρι τώρα ε, και τα 11 έχουν γίνει ήδη αποδεκτά για πιο μικρά ποσά στο πλαίσιο της ε, καταβολής ε, αυτής, των προκαταβολών 40 ε, εκατομμύρια. Θα πρέπει να δούμε αν το σύστημα των ε, προκαταβολών είναι αναλογικό και τι εμπόδια έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη για την καταβολή των σχετικών ετοιμάτων. Πραγματικά είναι πολύ πλοκή η διαδικασία, ε, για να πω το λιγότερο, της ε, υποβολής ε, αιτημάτων. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ε, ε, προϋποθέσεων να εκπληρώσουμε πρώτου μπορούμε να καταθέσουμε ένα αίτημα. Ε, αυτό πραγματικά δυσκολεύει πολύ τα πράγματα και για κάποιες διοικήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσω όλα αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει κατά πόσον θα μπορούσε να πλουστεύσει τα πράγματα Δεύτερον, αν είναι πράγματι κάτι που είναι ευκταίο, να έχουμε δηλαδή μια απλουστευμένη δικασία αποβολής ετοιμάτων για την κατάθεση των, ε, για την καταβολή προκαταβολής. Νομίζω ότι σε μερικέ περιπτώσει, ε, παραδείγματο χάρη, αν υπάρχουν πλημμύρε, ε, εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί αυτό. Δεν χρειάζεται να καταβάλλονται τόσα πολλά έγγραφα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο απλή και εύκολη για του ε, ετούντε η διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιο το λόγο. Αν όχι, θα πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι Είναι θεμελιώδες το θέμα. Θα ήθελα όμως να διαβουλευθώ με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ καταρχάς πριν μπορέσω να δώσω απάντηση. Γιατί πραγματικά το θέμα αφορά το όλο το, το, το επίκεντρο του πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Οπότε θα ήθελα αφού έχω τις ε, διαβουλεύσεις και συνομιλίες που πρέπει να επανέλθω σε σας γραπτός αν μου επιτρέπετε. Συμφωνείτε εσείς κυρία Χολμάιερ. Ωραία. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών είναι η 22 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Νοέμβριο θα λάβει χώρα. 21 συγκεκριμένα Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Πηγαίνουμε στο σημείο 13 που είναι ανταλλαγή απόψεων ε, σε σχέση με την κτηριακή πολιτική τη... και σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, στο της Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σεπτέμβριο στις 24 του μήνα είχα μια ανταλλαγή απόψεων για την κτηριακή πολιτική μαζί με την Κομισιόν. Τώρα θα συστήσουμε τη δική μας κτηριακή πολιτική. Με βάση το ετήσιο έγγραφο εργασία, καλωσορίζω στην Επιτροπή του δύο του Προέδρους που έχουν αρμοδιότητα ακριβώ στην κτηριακή πολιτική. Α, δεν μπορώ να του καλωσορίσω γιατί δεν είναι ακόμη εδώ. Άρα θα πρέπει να του περιμένουμε. Εκ νέου ολιγόλεπτη διακοπή, ελπίζω ολιγόλεπτη. So the latest information is that the... Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Κλάους Βέλε, όπου να είναι καταφθάνει. Όμως δεν είναι εδώ ακόμη δύο αντιπρόεδροι. Ο κύριος Βίλαντ και ο Πέτρο Σίλβα Περέιρα δηλαδή. Επομένως, Let's. Is somebody arriving or not? There. Can we start with him? I would say so. Yeah. Okay. Welcome. Please have a seat. Are you ready, Mr. Vella? I'm ready. Κύριε Βέλλε, είστε έτοιμος? Είμαι. Οπότε ξεκινούμε με τον κύριο Βέλλε. Έχετε το λόγο. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος ε, έχει πέσει σε κίνηση. Γι' αυτό μου ζητήθηκε να λάβω εγώ πρώτα το λόγο. Ευχαρίστω να το κάνω. Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για την κτηριακή πολιτική με βάση την έκθεση την οποία, την οποία καταθέσαμε στα τέλη προηγούμενη ε, κοινοβουλευτική θητεία. θητείας. Εισαγωγικά ίσως να πω ότι το 2010 Είχαμε την πρώτη μεσοπρόθεσμη κτηριακή στρατηγική. Στόχο τότε ήταν να έχουμε παρκή γραφεία για τη διάθεση των ευρωβουλευτών, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο της τελευταίας ε, θητείας νομίζω ότι καταφέραμε να αυξήσουμε κατά πολύ την έκταση. Το 2016 πήραμε τον Τεμέους, βέβαια με μίστομα, αλλά ε, η χίλιοι πάλι μπορούν να, να φιλοξενηθούν εκεί. Έχουμε την ανανέωση για την ε, επόμενη χρονιά, 2017, είχαμε το Ευρωπαϊκό Σπίτι της Ιστορίας που άνοιξε, το 2018 το Μάρτενς. Χίλιοι περίπου εργαζόμενοι και σίγουρα χαλάρωσε αυτό κάπως ε, το συνοστισμό η γάμα προσωπικού συνεργάζεται στενά μαζί μας ε, για να υπάρξει μεταφορά σε ένα κτίριο όλου του προσωπικού της και στα τέλη αυτού του έτους ε, θα ξεκινήσουμε και ε, την γέννηση στο Λουξεμβούργο. Γάμα και προβλέπεται και για τις άλλες γενικές διευθύνσεις πριν το καλοκαίρι. Το 70% δηλαδή της πρώτης φάσης ε, των δομικών έργων θα έχει κλείσει στο Λουξεμβούργο. Όλα αυτά τα κτίρια, όλα αυτά τα κτηριακά έργα τα έχουμε ε, εντάξει στον προπλησμό χωρίς κανένα κόστος, υπέρβασης κόστους. Έχει ολοκληρωθεί πλήρωση χρηματοδότηση, έχουν πληρωθεί δηλαδή και ό,τι άλλο προκύψει θα το καλύψουμε. Σε ό,τι αφορά αυτές τις δραστηριότητες και σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη τη στρατηγική του 2010, τον Απρίλιο ε, του 2018 ε, το Προεδρείο ψήφισε μία νέα κτηριακή πολιτική που βάζει κάποιους μεσοπρόθεσμους στόχους. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά ε, τη διάθεση γραφείων δεν είναι πλέον ο βασικός στόχος της κτηριακής ε, πολιτικής μας, διότι έχουμε ε, κατά το μάλλον ή τον επιτελέσει αυτό το στόχο για τους βουλευτές. Έχουμε ένα γραφείο συνδύο για τους βοηθούς στο Στρασβούργο. Μετά από 40 χρόνια για πρώτη φορά έχουμε ένα, ένα γραφείο για το βουλευτή και ένα ξεχωριστό για το βοηθό. έχασε 300 γραφεία η διοίκηση για να μπορέσει να τα διαθέσει στους βουλευτές. Με την εκτεριακη στρατηγική τώρα, Φεβρουάριο, Απρίλιος του 2018, ετέθησαν νέες προτεραιότητες για την κτηριακή στρατηγική που είναι πρώτον ανακαίνιση Έχουμε πλέον την ιδιοκτησία ε, κτηρίων πάνω από ένα εκατομμύριο τετραγωνικών ε, μέτρων ε, και το 3% το ανακαινίζουμε κάθε χρόνο. Αυτό, αυτή είναι η υποχρέωση, 3% των, της έκτασης ετησίως να ανακαινίζεται, που σημαίνει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρήσει τον κανόνα αυτό. Δηλαδή μέσα σε 33 έτη ουσιαστικά όλα τα κτίρια τα οποία είναι στην οικογένεια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχουν ανακαινιστεί. Έχουμε λοιπόν και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για να βλέπουμε περίπου πότε, ποια χρονιά και ποια κτίρια θα πρέπει να ανακαινίζονται. Δεύτερο στόχο σημαντικός ε, είναι ε, για την εμπειρία Ευρώπη ε, να επεκτείνουμε αυτό το έργο και στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και το τρίτο, ο τρίτο στόχος είναι να ε, βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις για τους ε, τριμερείς διαλόγους ε, διότι σε αυτά τα κτίρια δεν γίνονταν τριμερείς διάλογοι, αν γίνονταν ήταν σε πολύ περιορισμένη έκταση και για τις περισσότερες επιτροπές όμως εκεί συζητούνται ουσιαστικά ε, και αποφασίζονται τα διάφορα ζητήματα. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις ε, προτεραιότητές μας. Σε ό,τι αφορά τις ανακαινήσεις, ε, έχουμε το ΣΠΑΚ ως πρώτη προτεραιότητα. Εδώ το Προεδρείο αποφάσισε και στην ε, προηγούμενη ε, θητεία να ξεκινήσει έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα δώσει τη δυνατότητα το καλοκαίρι του 2020 στο Προεδρείο με βάση εναλλακτικών προτάσεων να λάβουν μια απόφαση για το πώς θα προχωρήσει η ανακαίνιση αυτή. Ε, πρέπει να γίνουν βέβαια οι αναλύσεις ε, οι σχετικές. Έχουμε ήδη κάνει αυτή τη διαδικασία και ε, ο διαγωνισμός ε, έχει λάβει υπόψη. Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο επιλογές, η ανακαίνιση ή ανακατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη οι αρχέ που θα συμμετάσχουν, δηλαδή να κατάσχουν πατάσει και για τι δύο εναλλακτικέ. Οπότε το Προεδρείο θα μπορέσει να αποφασίσει τα δέοντα. Έχουμε το πρωτόκολλο, την ασφάλεια ε, για τους τριμερείς διαλόγους και όπως είπα το Εμπειρία Ευρώπη. Αυτά είναι τα βασικά. Σε ό,τι αφορά το Experience Europe, ε, τους ε, μικρούς βουλευτές, επτά έχουμε αυτή τη στιγμή ή τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στην Κοπενχάγη, στο και στη Λιουμπλιάνα, στο Βερολίνο και στο Ταλίν και προβλέπονται ακόμη 7 για Λουξεμβούργο, Παρίσι, Ρώμη, Δουβλίνο, Στοκχόλμη, Βαρσοβία, Πράγα. Ώστε στα μισά κράτη-μέλη με βάση αυτό το προγραμματισμό στα τέλη της ε, θητείας ε, να έχουμε τέτοιες ε, εγκαταστάσεις. Το Προεδρείο σε μία ε, σύσκεψή του το μελέτησε ε, διεξοδικά το θέμα για να δούμε τι άλλες δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά στους τεμερείς διαλόγους, θέλουμε να είναι ασφαλή, 60 με 80 θέσεις, να είναι ασφαλής η χώρη αυτή και να μπορεί να παρέχεται ε, διερμηνία σε τουλάχιστον 6 γλώσσες για για τους βουλευτές. Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν, εμπειρία Ευρώπη, ανακοινήσεις και τριμερείς διάλογοι. Αυτά λοιπόν είναι στο σχεδιασμό μας ε, και σε αυτή την ε, θητεία αυτά είναι τα βασικά, αυτή είναι η βασική μας στόχη. Και φαντάζομαι ότι και με τη δική σας την Επιτροπή θα συζητήσουμε αναλυτικότερα οτιδήποτε ε, θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σιλό Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερο που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όπως ε, θα γνωρίζετε, είμαι ο αρμόδιος αντιπρόεδρος για τα κτίρια. Α, αλλά ω δεύτερος αντιπρόεδρος για τα θέματα αυτά, ο πρώτος αντιπρόεδρος για θέματα και πολιτική είναι ο κύριος Βίλαντ. Γι' αυτό και περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση και προσβλέπω σε γόνιμη συνεργασία με την Επιτροπή. Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε το έγγραφο εργασία του 2019 με θέμα την κτηριακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για το υπόβαθρο αυτού του εγγράφου και να σας αναλύσω κάπως την νομική βάση που διέπει τις σχέσεις μας. Γιατί γνωρίζω ότι για πολλούς ευρωβουλευτές όλα αυτά είναι καινούρια. Γιατί πολλοί είναι νεοκλεγέντες. Θα σας πω λοιπόν δύο λόγια για το πού βρισκόμαστε μετά την διεξοδική παρουσίαση που μας έκανε ο Γενικός μας Γραμματέας. Το κύριο στοιχείο της κτηριακής στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μία απόφαση του 1992 που προέβλεπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εστιαστεί στην αγορά των ακινήτων του. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είμαστε ιδιοκτήτες το 80% των κτηρίων που χρησιμοποιούμε. Αυτή η εξέλιξη είναι θετική κατά τη γνώμη μας, γιατί χάρη σε αυτή την αγορά εξοικονομήσαμε πολλά κονδύλια από μισθώματα. Βέβαια έχουμε άλλα έξοδα, όπως είναι η, ανα... η η συντήρηση όλων αυτών των κτίριων, στα οποία έχουμε την κυριότητα. Το 2010 εκπονήσαμε την πρώτη μέσο και μακροπρόθεσμη κτηριακή μας πολιτική και στη συνέχεια, το 2018, είχαμε το νέο στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το μέλλον, δηλαδή μετά το 2019. Με βάση τις προτεραιότητες μας, ε, τις προτεραιότητες που είχαμε τότε, η μέρη μας είναι να προσαρμόσουμε τις εγκαταστάσεις μας ε, στις ε, εξελίξεις, τις αλλαγές σε ό,τι αφορά τα Τη έδωση συνεδρίασης ώστε να λαμβάνουν υπόψη και του ε, τριμερεί διαλόγου. Επίση, ε, έχουμε στα γραφεία συνδέσμου το mainstreaming του Εμπειρία Ευρώπη. Επίση είχαμε την εσωτερική ανάθεση τη ασφάλεια των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ανάγκη εξασφάλιση διασύνδεση των κεντρικών με κτηρίων. Η ανακαίνιση των κτηρίων μα. φυσικά εξακολουθεί να είναι σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε Βέβαια, από αυτήν την άποψη έχουμε σημαντικές βελτιώσεις της κατάστασης. Ιδιαίτερα έχουν βελτιωθεί οι εργασιακές συνθήκες και για τους ευρωβουλευτές και για τους υπαλλήλου. και κάθε ευρωβουλευτή έχει πλέον περισσότερα γραφεία στη διάθεσή του. Επίσης έχουμε ε, μια πιο μοντέρνα διαρρύθμιση των ε, γραφείων και γενικώ οι, οι χώροι είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες. Mm. εξυγχρονίσαμε ταυτόχρονα και τις υποδομές μας και το, την επίπλωση και τον εξοπλισμό των γραφείων. Επίσης είχαμε αισθητέ ε, βελτιώσεις και στο μπαρ στο Στρασβούργο και στο lounge εδώ στις Βρυξέλλες και στα εστιατόρια. Lounge. Επίσης ε, και στο Κισμέλο θα έχουμε ένα νέο Lounge και βελτιώσει έγιναν και στα γραφεία συνδέσμου, κυρίως με το Εμπειρία Ευρώπη και φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε το Παρλαμεντάριο και τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Επίσης, ανακαινήσαμε και κτίρια μας στο Λουξεμβούργο και κυρίως ε, το σύμπλεγμα κτιριών Κόνραντ Αντενάουερ. Βέβαια έχουμε αρκετές προκλήσεις στο μέλλον. Έχουμε την ανακαίνιση, την επικείμενη του κτίριου Polaris Park. Επίσης, τι θα γίνει με το παλιό κτίριο Denauer, που δεν θα μας χρειάζεται πια. Τουλάχιστον όχι με την ίδια ένταση που το χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν. Επίσης, υπάρχει πρόθεση να επεκτείνουμε αυτή την εμπειρία Ευρώπη στα γραφεία συνδέσμου. Θα έχουμε τι νέες εγκαταστάσει για τους επισκέπτες στο νέο κτίριο που, που περνάει πια στη δεύτερη φάση. Επίσης έχουμε την συζήτηση για το πώς θα πρέπει να γίνει εσωτερική ανάθεση των πόρων διαχείρισης για τα διάφορα γραφεία συντήρησης και θέλουμε να βελτιώσουμε και τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, υιοθετώντα πιο φιλόδοξους στόχους. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία τώρα που έχουμε για τη διαχείριση των κτηρίων μας, η διαχείριση φυσικά των κτιρίων διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό και με βάση τον δημοσιονομικό κανονισμό κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, παρέχει στην, θα παράσχει στην ε, αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή ένα έγγραφο εργασίας με θέμα την κτηριακή του πολιτική. Όπως και έγινε με το έγγραφο που εκπώνησε το προηγούμενο Προεδρείο για την κτηριακή πολιτική για το 2019. Επίσης, βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού, για κάθε σχέδιο ε, για νέο κτίριο που θα έχει σημαντικέ δημοσιονομικέ συνέπειε. το αρμόδιο θεσμικό όργανο θα πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό. Οπότε κάποια σχέδια θα πρέπει να κοινοποιηθούν εγκαίρως στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης. Γιατί προϋποθέτει κάποια προέγκριση. Επίση, τα σχέδια αυτά που εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία τη έγκαιρη ενημέρωση συνήθω υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω αυτού του εγγράφου εργασία για την κτηριακή πολιτική, αλλά μπορεί να υποβάλλονται και στην Επιτροπή Προπολογισμών με άλλη βάση. Βέβαια, αποτελείται προέγκριση για όταν χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις για επιμέρους σχέδια. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο εργασίας του 2019, δόθηκε έγκαιρη ενημέρωση, ιδιαίτερα για τα γραφεία συνδέσμου. Εκεί παρέχονται πληροφορίες για την Πράγα, Βαρσοβία και Στοκχόλμη, για τα τρία γραφεία συνδέσμου στην Πράγα, Βαρσοβία και Στοκχόλμη. Δίνονται πληροφορίες λοιπόν για αυτά τα γραφεία στη και για την ε, εγκατάσταση του Εμπειρία Ευρώπη. Επίσης δόθηκε εμπρόθεσμη ενημέρωση για τον εξοπλισμό ε, του εστιατορίου εδώ των Ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες. Εκεί έχουν γίνει σχέδια για σημαντική ανακαίνιση. Βέβαια θα μειωθεί ο αριθμός των θέσεων στο εστιατόριο, αλλά θα αυξηθούν τα ε, σαλόνια σε 10 θα διπλασιαστούν δηλαδή υπάρχουν, τα υπάρχοντα. Και συνεχίζουμε τον εξοπλισμό, την ε, ανακαίνιση της επίπλωσης του μπαρ. Στο κτίριο αυτό το ASP. Αυτά σε γενικές γραμμές και είμαι πρόθυμος για την συζήτηση που θα ακολουθήσει και την ανταλλαγή απόψεων, στην προσβλέπω. Έρχεται ο κύριος Βίλαντα από ό,τι μου λένε, αλλά σας προτείνω να συνεχίζουμε με ναι, τις εργασίες μας, οπότε για τώρα θα σου το λόγο στην μόνιμη εισηγήτρια για την κτηριακή πολιτική, την κυρία Κέλλερ. Merci euh, beaucoup pour... Ευχαριστώ πολύ κύριε Κελέρη για αυτή σας την παρουσίαση κύριε Γενική Γραμματέα και κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής κύριε Βέλε και Περέιρα για όσα μας υποθυμίσατε για το πλαίσιο της κατάστασης. Βέβαια τα πράγματα κάπως ε, ιδιαίτερα είναι τα δικά μας κτίρια, τα κτίρια όπου εργαζόμαστε, τα κτίρια για τους ε, υπαλλήλους, τους βουλευτές και για όλους τους συνεργάτες ε, και γενικότερα το προσωπικό των πολιτικών ομάδων μας υπενθυμίσατε, το ιστορικό πλαίσιο και οι δύο. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο και σε ευχαριστούμε επίσης για αυτό το έγγραφο που μας έχετε διαβιβάσει, να το δείξω στην κάμερα. Και εκεί μας υπενθυμίζετε τα βασικά στοιχεία γιατί όντως δεν είναι πολύ εύκολο να δούμε τι γίνεται με το κάθε κτίριο. Και όπως είπατε κύριε Βέλεχτε, πρόκειται για ε, το κτίριο Paul Henry Spack και όχι PHS. Γιατί PHS είναι μια χημική ουσία, ένα προϊόν τέλος πάντων. Τώρα, έχω κάποιες ερωτήσεις. Ίσως είναι αυτό λίγο πρόβλημα στην αρχή της θητείας, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για την έκθεση για αυτό το κτίριο, το Polar Henry Σπάκ Είναι το θέμα. Σημαντικό και αναφέρατε κύριε Γενικέ ότι έχει γίνει αυτός ο διαγωνισμός για αρχιτέκτονα. Πρόκειται να δημοσιευθεί η πρόσκληση συντόμω για να δούμε κατά πόσο θα έχουμε ανακαίνιση ή μερική επανοικοδόμηση. Άρα για αυτό το θέμα μήπως πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους έγκαιρη πρώιμη προειδοποίηση ούτως ώστε να μπορούμε τα λογογνώσεις να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις αφού γνωρίζουμε τα θέματα και να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου. Λοιπόν, θα κάνουμε, θα χτίσουμε ή θα γκρεμίσουμε για να ξαναχτίσουμε για να ξέρουμε επομένως λαμβάνοντας τι υπόψη θα αποφασίσουμε σχετικά και εδώ είναι θέμα πολλών εκατομμύριων ευρώ άρα προσοχή αυτή τη φορά μας είπατε για το Λουξεμβούργο ότι υπάρχουν και εκεί σημαντικά έργα που προβλέπονται για το Αντενάουερ 2. Και εκεί, συνάδελφοι και υποφαινόμενοι, θέλουμε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά το συνολικό κόστος για το κτίριο. Επίσης το χρονοδιάγραμμα, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Επίσης, τρεις πόλεις για θεσμικό όργανο, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο και δεν ε, είδα να υπάρχει κάποια πρόταση για κάποια έργα, για κάποια επέκταση και από ό,τι κατάλαβα για την Ολομέλεια ότι υπάρχει ε, δυσκολία τόσο ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε εκεί κάποιες διοικητικές ε, υπηρεσίε και εξού και τα open space. Άρα αυτό θα μας παρουσιάσετε σύντομα και ε, αυτή τη μνήμα του 3%. 3% της αναγκαίας ετησίας επενδύσεως. Ως ε, κανόνα, ως ε, θεωρία αρχή χρηστής διαχείρισης για το Στρασβούργο. για την ευρωπαϊκή εμπειρία, Europa Experience. Αυτό ενδιαφέρει πολύ τους αδέλφους. Να δούμε πώς οι νέοι και λιγότερο νέοι ε, συμπολίτε μας να μπορούν να, να αποκτήσουν μια εμπειρία από το κοινοβούλιο, οπότε κάποια στιγμή και αυτό να μας το παρουσιάσετε. Τι γίνεται με όλα αυτά τα έργα και ε, και την εμπειρία σα από το παρελθόν. Πάντως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ε, αν θέλουμε να δούμε ε, κάτι σαν προσωμείωση ας πούμε το τι μπορεί να κάνουμε αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή υπόθεση. Αυτά για το σημαντικό αυτό ζήτημα και συμπαθάτε με κάτι είπαμε που τα γνωρίζετε καλύτερα από όλους, αλλά ε, αρχή της θητείας είναι. Εξού και οι πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Στο μεταξύ, ήρθε ο κύριος Βίλαν, καλώς ορίσατε. Και ας δώσουμε και σε εκείνον τώρα τον λόγο για μια εισήγηση. Οκτώ λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ähm. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σητώ συγγνώμη αλλά η κατάσταση ε, με την κίνηση με έκανε να καθυστερήσω. Δεν χρειάζομαι 8 λεπτά, αλλά λίγο προς τα πίσω να σας πάω και να πω ότι η κτηριακή πολιτική ήταν να, ε, είμαστε, να έχουμε στην κατοχή μας τα κτίρια και όχι να νοικιάζουμε. Αυτή ήταν η προτεραιότητα από πολιτικής πλευράς και βάσει αυτής κινηθήκαμε. Δεύτερον, η εσωτερικοποίηση, η εσωτερήκευση ε, και της ασφάλειας ε, και των ε, οδηγών ήταν κάτι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, αλλά νομίζω ότι εστέφθη με επιτυχία, την οποία θέλουμε να εδραιώσουμε. Και το τρίτο είναι κάτι επίμαχο, τα έπιπλα. Και νομίζω ότι και εδώ βλέπουμε την αρχή μιας επιτυχίας, μιας επιτυχούς προσέγγισης Και βέβαια υπάρχει ε, η ανάγκη να λάβουμε ε, διάφορα κριτήρια υπόψη. Έχουμε τώρα και την ανακαίνιση που ε, πρέπει να λάβει υπόψη το Brexit, βέβαια, το ότι δεν θα έχουμε τους Βρετανούς βουλευτές μαζί μας. Αλλά προς το παρόν είναι ανοιχτά τα πράγματα, πιο, για πιο πολύ διάστημα από ό,τι περιμέναμε. Έχουμε κάνει πιλωτικά προγράμματα ε, με πέντε συναδέλφους και έχουμε πλέον ανοίξει νέες ε, άγουσες, οποίες θα διερευνήσουμε και στο μέλλον. Θέλω να πω επίσης ότι το, η μεγαλύτερη πρόκληση, το μεγαλύτερο εργοτάξιο αν θέλετε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι το PHS και ο γενικός ε, γραμματέας φαντάζομαι ότι σας ε, το είπε. Αν δεν έχετε ενημερωθεί αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε νέοι, ε, παρακαλώ να δείτε τι ε, λέει και στην ισοσελίδα της η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ η αρμόδια γιατί με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο PHS, στο Polonary SPAC, έχουμε τα προβλήματα της ασφάλειας. Όσο δεν τα έχουμε εντελώς ε, λύσει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε στο Προεδρείο, διότι δεν έχουμε ακόμη εντελώς αποφύγει προβλήματα για το Εμπειρία Ευρώπη, είπατε και εσείς ε, κυρία Κελέρα, εγώ είμαι φίλος αυτής της πρωτοβουλίας και νομίζω ότι πρέπει να την ε, προωθήσουμε ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να βρούμε έναν ε, άλλο τρόπο συνεννόησης, ένα μόντους βιβέντη με την Επιτροπή, με τον κύριο Έτιγκερ τα είχαμε βρει κατά κάποιο τρόπο και με τον Επίτροπο Χάν πιστεύω, επί Παρίσι Δουβλίνο για διάφορους λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο πολύ με του σπόρους, αλλά δεν είχαμε σίγουρα και την επαρκή χρηματοδότηση που εμείς θα θέλαμε. Είχαμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τώρα με την απόφαση αγορά ή μίσθωμα ε, την έκταση, την επιφάνεια και όλα αυτά, τώρα πρέπει να ε, συνεργαστούμε σε νέε βάσει εντελώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σα μιλάω για το Παρίσι και για τη Ρώμη και για το Δουβλίνο, που επειδή είναι και τελείω διαφορετικέ οι αγορέ, Υπάρχουν κάποιοι εταίροι που πρέπει να λάβουν υπόψη και νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν θα προβούμε σε μια αλλαγή παραδείγματος. Μήπως θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ νωρίτερα τις σχετικές αποφάσεις για να μπορούν να ξεκινούν πάρα πολύ νωρίτερα οι διαδικασίες με την εκμίσθωση των κτηρίων. Σε μια σύσκεψη του Προεδρείου το είπα και για τα έπιπλα με κάποιες ε, ιδέες οι οποίες ακούστηκαν, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική. Ε, χρειάζεται ένας προβληματισμός, ε, να έχουμε αν θέλετε ένα εργαστήριο ανταλλαγή απόψεων προβληματισμού. χρειάζεται ένα εργαστήριο ώστε από νωρίς να μπορούμε να δοκιμάζουμε κάποιες ιδέες, να δούμε τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, ε, παραδείγματο χάρη προτάσεις μπορούμε να καταθέσουμε στην αθέλφους για να μπορούν να τις ε, μελετήσουν. Έχουμε κάποια ακουάριου, τα λέω εγώ, κάποια ενιδρία. Είναι τα, κάπως ε, σαν ενιδρία την είναι όλο με γυαλί. Υπάρχει το ε, online booking, μπορούν και οι βουλευτές ε, online να κλείνουν αυτές τις αίθουσες ε, σύσκεψης έχουν ε, αυξηθεί. Θέλω να έχουμε μια δεξαμενή πόρων για την κατανομή των κρατήσεων και ο καθένας με τις δυνατότητές του να μπορεί να συμμετέχει. Νομίζω ότι είναι οι συνέργειες πάρα πολλές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εγγραφή στον προϋπολογισμό, ιδίως για τις επιτροπές. Έχουμε κονδύλια για τις επιτροπές από καφέ ε, μέχρι τα ταξίδια των αντιπροσωπιών και τα χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά τελείως διαφορετικά οι διάφορες ε, επιτροπές. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι Παραδείγματο χάρη, όταν ακυρώνονται τελευταία στιγμή κάποιε συνεδριάσει, τι γίνεται με τη χωρητικότητα των συνεδριάσεων, πόσε γλώσσε, δηλαδή πόσοι διερμηνεί χρειάζονται. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν ξέρω, ίσως να προσφέρετε λιγότερο καφέ και να μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε κάποια ταξίδια αντιπροσωπιών με πιο επαρκή προϋπολογισμό ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε καλύτερα τώρα των επιτροπών, αλλά να εξοικονομούμε ή τέλο πάντων να μπορούμε να διχειριζόμαστε με πιο οικονομικό τρόπο του σπόρου που έχουμε στην ε, ε, διάθεσή μα. Παραδείγματο χάρη, μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα να μπορούν να γίνονται συνεδριάσει, γιατί έχουμε κάποια συγκεκριμένα κτίρια, κάποιε συγκεκριμένε εκτάσει μπορούμε να διαθέσουμε και βλέπουμε ότι πέφτουν όλοι, όλε οι συνεδριάσει σε λίγε ε, ώρες εχμής και ημέρες εχμής την εβδομάδα και καλό θα ήταν να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασπορά. Ε, νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει και τις ίδιες τις ε, επιτροπές. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επανέρχομαι τώρα στους συναδέλφους. Κυρία Χολμαέρ. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω απόλυτα τα όσα είπε η κυρία Κέλλερ σε ό,τι αφορά το PHS, ε, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να βρούμε μια λύση, το Poland Pack. Ίσως ε, ανακατασκευή για να μπορεί να μας εξασφαλίσει ε, την ασφάλεια, διότι αυτά που έχω διαβάσει πραγματικά δεν με ικανοποιούν και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Γιατί δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο είναι ανακαίνιση επαρκή. Δεύτερον, για το σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μάλλον το House of Europe ε, στο Βερολίνο και αλλού πρέπει να ε, προωθήσουμε ε, τα γραφεία αυτά να είναι ένα σημείο αναφοράς για τους πολίτες. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στους πολίτες των χωρών. Κάποιοι δεν θέλουν ε, σε κάποια κράτη-μέλη τόσο πολύ να προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα αυτό δεν είναι θετικό. Επομένως ε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί στο δυνατό περισσότερος κόσμος να επισκέφτεται αυτά τα γραμμία, γραφεία και να έρχεται σε επαφή ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Παρίσι νομίζω υπήρξαν ε, κάποιες ε, προτάσεις ε, να μετακινηθεί το γραφείο σε ένα σημείο που μπορεί να μην είναι τόσο δαπανηρό, αλλά δεν θα πηγαίνει κανείς εκεί. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο φθηνό το Παρίσι τώρα, όχι τόσο δεν έχει ακριβή, είναι, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα έπιπλα, νομίζω βρέθηκε μια καλή λύση ε, να μην αγοράζουμε αλλά να μισθώνουμε είναι ένα καλό μοντέλο. Έχουμε πάνω από 700 βουλευτές ε, και υπάρχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες ε, για τη χρήση των επίπλων. Νομίζω λοιπόν ότι η λύση που βρήκατε είναι η βέλτιστη δυνατή. Αυτές, αυτά τα, η θάλαμη αυτή από γυαλί επίσης είναι μια πολύ θετική ιδέα μικρές δομές είναι κάτι το οποίο είναι μια προσέγγιση που ακολουθείται, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Θέλουμε πολυλειτουργικούς ε, χώρους σήμερα. Αλλά καμιά φορά η τεχνολογία δεν έχει προωθηθεί τόσο πολύ και Στο ό,τι αφορά τα δικά μου γραφεία, έχω ε, πολυλειτουργικά κουμπιά μόνο, αλλά δεν είναι και τόσο. Πολυλειτουργικού πολυλειτουργικούς ε, εκ, εκτυπωτές, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για το οτιδήποτε. Ε, Είναι πράγματι κάτι πολύ χρήσιμο αυτή η λειτουργική εκτυπωτέσα του συστήνω. Επομένως όπου έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία ε, νομίζω ότι είναι καλό γιατί οι εκτυπωτές χωρίς ε, πολυλειτουργικά κουμπιά και δυνατότητες λειτουργικές ε, δεν είναι normal, πώς να το πω ε, δεν θα το έπαιρνα ούτε και στο σπίτι μου ένα τέτοιο εκτυπώτη. Πραγματικά θέλω να ε, το επενέσω αυτό, τον σύγχρονο εξοπλισμό. Πραγματικά έχω ανανεωθεί ε, επίσης. Δεν είναι όλα πια γκρι, είπα και τα έπιπλα είναι πολύ ευχάριστα. Νιώθω πολύ έτσι ευχάριστα ε, σε σχέση με πιο παλιούς καιρούς ε, και αν προωθηθεί η τεχνολογία, βελτιωθεί και σε κάποια πράγματα ακόμη, ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο χαρούμενη θα είμαι. Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόσακοφ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. Έχω περισσότερε ερωτήσει παρά σχόλια, γιατί είμαι νέο ευρωβουλευτή. Καταρχήν για το πω, κτίριο Polar πακ. Βλέπω δύο αριθμούς εδώ. Ε, 400.000 είναι η εκτίμηση για, την ανακαίνιση, ενώ ήταν 500 εκατομμύρια το κόστος ανα, ανοικοδόμησης. Κάποιο λάθος, κάποιο λάκκο έχει φαμπαδό. Είτε είναι πολύ μικρό το ένα ποσό, είτε πολύ μεγάλο το άλλο. Θα ήθελα όταν υποβάλλεται συγκεκριμένα ποσά και εκτιμήσεις να είναι τεκμηριωμένα ώστε να μπορούμε και εμείς εμπεριστατωμένα να κάνουμε την επιλογή μας. Επίσης, τι γίνεται με τις σύραγγες που συνδέουν τα διάφορα κτίρια της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. έχει νόημα να χρηματοδοτήσουμε τέτοια έργα, μια και ήδη ο προπολογισμό μα είναι τσιμα-τσιμα. Επίση, για την ασφάλεια. Οι εγκαταστάσει και τα κτίρια είτε θα είναι ασφαλή είτε όχι ασφαλή. Αν δεν είναι ασφαλή θα πρέπει να το διορθώσουμε και να τα θωρακίσουμε το συντομότερο το δυνατό. Και επίση να δούμε τι περιορισμού έχουμε και τι χρονικού περιορισμού. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ασφάλεια στου δημόσιου χώρου, είναι κάπω προβλήμα προβληματικό. Και δεν είναι μόνο για τους ευρωβουλευτέ όταν λέμε για την ασφάλεια, αλλά και για όλο το προσωπικό, για όλου του υπαλλήλου. Επίση, θα ήθελα να κάνουμε κάποιες οργανωμένες ε, ε και να μας δείξετε επιτόπου τι σχεδιάζεται. Έτσι θα είναι και παιδαγωγικό και χρήσιμο και έτσι θα μπορέσουμε πιο περιστατωμένα και με πιο επαγγελματικό τρόπο να κάνουμε τις επιλογές μας. Μπορείτε λοιπόν να μας ξεναγήσετε σε όλα αυτά τα σχέδια που θα κάνετε. Ο κύριος Ανδρίασεν. Εγώ ακόμη είμαι σε φάση εξοικείωσης και εκμάθησης. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω όλα αυτά τα θέματα διεξοδικά. Εγώ έχω μια ερώτηση για την ενεργειακή απόδοση των κτίριων, γιατί έχουμε τεράστια πρόκληση με το κόστος της ενέργειας. Και όταν μιλούμε για το κλίμα, για τις κλιματικές αλλαγές και βλέπουμε τις τάξεις μεγέθους, θα πρέπει και εμείς να εντείνουμε τις προσπαθίες μας και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτίριων μας. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ενημερωτικά δύο λόγια για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Πολλές ε, ε, ερωτήσεις συγκεκριμένες και πολλά σχόλια έγιναν. Οπότε περιμένουμε τις απαντήσεις των τριών καλεσμένων μας εδώ, των δύο αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέως. Θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά με προηγουμένω. Οπότε πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Βέλε. Äh, Σα ευχαριστώ πολύ για την κυρία Κέλλερ καταρχά, για το ΣΠΑΚ. ισχύουν ε, οι αποφάσεις τελευταίας ε, θητείας, ε, ενημέρωση, early warning. Αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον, ώστε και η μόνιμη συγκήτρια αλλά και η Επιτροπή Προϋπολογισμών να ενημερώνονται σταθερά και διαρκώς για τις εξελίξεις αυτό το φάκελο. Να υπάρχει δηλαδή πλήρη, συνεχής ροή πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά το Αντενάουερ, η Επιτροπή Προπολογισμών Έχουμε τα, 4, 432 εκατομμύρια ε, Αυτό εγκρίθηκε από την ε, Επιτροπή Προπολογισμών ε, σε σταθερές τιμές. Αυτό είναι το κόστος. Σε ό,τι αφορά τώρα το Προεδρείο ασχολήθηκε με αυτό το project και πριν το τέλος της θητείας και σε ό,τι αφορά αυτό το ποσό Είμαστε κάτω του ορίου κατά 12,4 εκατομμύρια. Αν ε, ληφθούν υπόψη ε, τα άλλα έξοδα, έξοδα χρηματοδότησης, είμαστε και με αρκετό περιθώριο ασφάλειας 32,9 εκατομμύρια κάτω από το εκτιμόμενο ποσό. Γιατί το κόστος χρηματοδότησης είναι χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που περιμέναμε και γιατί λάβαμε υπόψη και χρησιμοποιήσαμε τα ε, πλεονάσματα τα οποία είχαμε και τα χρησιμοποιήσαμε. Άρα ε, όλα πάνε βάση του σχεδίου μέχρι τώρα. Η πρώτη τώρα ε, σειρά για το αντενάωρ των προσφορών ήταν πάνω από την εκτίμηση του κόστους, γύρω στο 1 τρίτο πιο πάνω και αποφάσισε το Προεδρείο να προκηρύχθει νέος διαγωνισμός, να μην δεχθούμε τις προσφορές δηλαδή που είχαμε λάβει. Έχουμε λοιπόν ε, μία νέα ε, πρόσκληση υποβολής προσφορών, άρα έχουμε πιο φθηνές προσφορές, όμως σίγουρα χάσαμε χρόνο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καθυστέρηση. Όποιοι ξέρετε τα μεγάλα κλιμακά κτηριακά έργα, Συνήθω έχουμε τρει ε, μεταβλητέ ε, ε, ποιότητα, τιμή, διάρκεια. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε κακή ποιότητα ούτε φθηνή τιμή ως προτεραιότητα, γι' αυτό καθυστερούμε λίγο. Σε ό,τι αφορά το Στρασβούργο υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο της προηγούμενης θητείας, Πήραμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης πλήρως ανακαινισμένο κτίριο, ε, το Χάβελ, το κτίριο Χάβελ. Επίσης, όπως ε, βλέπετε και στο έγγραφο, κάθε βουλευτής έχει ένα γραφείο δικό του συν ένα ακόμη. Στην προηγούμενη θητεία, επίσης, οικοδόμησαμε το ε, Εμπειρία Ευρώπη, κάτι πολύ ε, θετικό. Δύο εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση για την για το ΣΥΡΜΕΚ, το Memorial και στον τομέα της ασφάλειας ε, πολλές επενδύσεις ακόμη. Και θέλουμε να επενδύσουμε ε, στην είσοδο Λόου με ένα ε, ξεχωριστό κτίριο 2 εκατομμύρια ευρώ θα είναι μάλλον το κόστος, έχει σχεδιαστεί, εγκριθεί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το έργο και στο ΒΙΚ ε, η καντίνα πρέπει να ανακοινιστεί. Άρα και στο Στρασβούργο υπάρχουν έργα τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Για τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο προσπαθούμε ταυτόχρονα να προχωράμε, παράλληλα τις εργασίες, όχι μόνο πρώτα το ένα μετά το άλλο, αλλά ε, εκτιμώντας και την ανάγκη, τις ανάγκες επιτόπου να προσπαθούμε να προχωρούμε παράλληλα. Έχουμε μια ειδική κατάσταση τώρα, ιδιαίτερη κατάσταση στο Στρασβούργο μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχές του έτους, ε, είχαμε προγραμματίσει για 725 και όχι για 751 βουλευτές. Υπάρχουν τα γραφεία τα οποία πρέπει να κατέχουν ακόμη και θα μείνουν και κάποια κενά γραφεία στη συνέχεια. Έρχονται βέβαια κάποιοι ε, επιπλέον, αλλά δεν θα είναι σίγουρα 50 τον αριθμό. Θα είναι λιγότεροι, οπότε έχουμε ένα περιθώριο σε ό,τι αφορά την ε, χωρητικότητα. για του εκπροσώπους των κρατών μελών που παρίστανται τακτικά στο Στρασβούργο για το Experience Europe. Επίση, ε, θα σας ενημερώνω σας είπα ότι έχουμε 7 και άλλα 7 ε, τα προγραμματίζουμε, δηλαδή τα μισά στο πλαίσιο αυτής της θητείας, τα μισά κράτη μελή, την κυρία Χολμάιερ, το Experience Europe. Πράγματι θα είναι επιτυχή αν πηγαίνει κόσμος εκεί. Ε, είμαστε νομίζω επιτυχημένοι κατά το παρελθόν στο Ελισίνκι. 100.000 επισκέψεις σε λίγους μήνες γιατί είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Οπότε υπάρχουν πολλοί εκεί και μπορούν να πάνε να επισκεφθούν και αυτό το, το χώρο. Για το Βερολίνο 150.000 ε, είναι κοντά στο μνημείο του Μπραντ, αλλά γενικώ ε, πρέπει πράγματι να παροτρύνουμε και τα άλλα κρατημέλη να βρουν ε, χώρους που θα είναι κοντά ε, πολλοί κόσμος ή τέλος πάντων θα προσελκύουν κόσμο για να υπάρχει προσέλευση. Υπάρχει μια απόφαση του Προεδρού παλαιότερη που λέει ένα. Ε, στον εξοπλισμό, αλλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε σε ό,τι αφορά ε, Τώρα για το PHS, θα, σας τα είπα, ε, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις 380 εκατομμύρια αν γίνει πλήρης ανακατασκευή, αλλά εάν όλα αλλάξουν, πλην των θεμελίων 340 εκατομμύρια, άρα δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, θέλουμε όμως να δούμε και την τιμή, τις προσφορές που θα έχουμε. Δηλαδή να δούμε όχι μόνο πώς, αλλά και με τι τιμή θα προχωρήσουμε για να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο, μια πιο καλή εικόνα. Αλλά βλέπετε ότι η εκτιμόμενη ε, τιμή για τη μία ή την άλλη περίπτωση είναι κοντινές οι δύο, δηλαδή μια την αλλη περιπτωση ειναι κοντινες οι δυο δηλαδη μια διαφορα στα 10-15% μεταξύ ανακαίνησης ή ανακατασκευής και σε ό,τι αφορά την ε, γέφυρες τη διασύνδεση με την Κομισιόν για τούνελ δεν υπάρχει προβλέψη αλλά για ένα, μια γέφυρα. Υπάρχει μια συμφωνία με την περιφέρεια και με τους σιδηροδρόμους αλλά θα πρέπει να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας. Οι αρμόδιε δηλαδή υπηρεσίε της ΓΔ ΙΝΛΟ θα συμμετάσχουν, θα γίνει μια μελέτη, τεχνική μελέτη για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η γέφυρα και οι βελικές αρχές να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Να μπορεί κανείς πεζί με ποδήλατο ε, να πηγαίνει και να υπάρχει αυτή η σύνδεση για το Κοινοβούλιο όπως ε, με την Επιτροπή για το Συμβούλιο. Οπότε δεν θα είναι αποκομμένα μεταξύ τους τα όργανα, τα κτίρια τους δηλαδή. Το άλλο ερώτημα ήταν για την ενέργεια. Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλουμε ε, την καλύτερη ποιότητα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, το BREAM, αυτή η πιστοποίηση BREAM ε, και για το Adenauer το ίδιο θέλουμε. με βάση τα τελευταία περιβαλλοντικά και ενεργειακά πρότυπα θέλουμε να κατασκευάζουμε. Πρέπει να βλέπουμε όμως ε, και τι ε, ενεργειακή απόδοση έχουν τα κτίρια μας και αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση ή εξυγχρονισμό. 2024 θέλουμε στο Κοινοβούλιο να έχουμε ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, έχουμε την διάμεση φάση με υβριδικά αλλά η περιβαλλοντική στρατηγική την οποία αποφάσισε το Πρόεδρο αυτό προβλέπει. Είμαστε πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό. Και θέλουμε κατά 95% επίσης πράσινες δημόσιες προμήθειες. Αυτό είναι συστηματική πολιτική λοιπόν ε, της, ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος ε, από τους δύο κυρίους. Πρώτον, να σας πω ότι έξι ώρες πρέπει να σταματήσουμε γιατί δεν θα έχουμε πλέον διερμηνία. Πρέπει να αποχωρήσουν οι διερμηνείς. Κύριε Βίλαντ, έχετε εσείς το λόγο. Είναι πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Στάκοφ, ε, νομίζω τα απάντησε για το κόστος ε, ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί εγώ με τη διοίκηση ίσως να μην είμαι 100% σύμφωνος για το άτριουμ, για παράδειγμα. Για τους ε, επισκέπτες. Οι ομάδες επισκεπτών, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να, να πηγαίνουν στο άτριουμ. Ε, μετά μπορεί να θέλουν να πάνε στο ημικύκλιο, να βγουν, να ξαναμπούν. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε με αρχιτεκτονικό ε, διαγωνισμό. Υπάρχουν κάποια σημεία διαπαφής ε, με το άτριουμ. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να μεταφέρει τους ε, επισκεπτές από το άτριουμ στην αίθουσα του ημικυκλίου χωρίς να περνάνε δύο φορές έλεγχο ασφαλείας, για παράδειγμα. Ένα άλλο. στο άσπα Έχουμε δύο εκατομμύρια γεύματα. Τι γίνεται με τους ε, μάγειρους. Ε, ε μήπως ε, θα πρέπει να υπάρχει μία κουζίνα. αν χρειαστεί να δημιουργηθεί νέα και να ανακαινηθεί η κουζίνα στο ΑΕΣΠΕ, πώς θα ανακαινήσουμε ε, μια κουζίνα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχονται τα γεύματα, να εξασφαλίζεται η παροχή γευμάτων. Νομίζω σε ό,τι αφορά το, τους ανελκυστήρες δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά είμαστε σε συνεχή επαφή με τους κατασκευαστές για την ευφυή καθαριότητα. Ε, επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το δούμε γιατί κοστίζει σε προσωπικό, κοστίζει σε ενέργεια Παραδείγματο χάρη, όταν είμαστε στο Στρασβούργο, δεν χρειάζεται να καθαρίζονται εδώ τα ε, γραφεία στι Βρυξέλλε. Υπάρχουν τεχνολογίε ε, με τι οποίε μπορούμε με έναν υπολογιστή να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην υιοθετήσουμε πάρα πολύ προχωρημένες τεχνολογίες που ε, όταν τις σχεδιάζουμε δηλαδή είναι πάρα πολύ προχωρημένες, αλλά μέχρι να χρησιμοποιηθούν ήδη είναι ξεπερασμένες. Και για τους εκτυπωτές ήταν στην Ίνλο. Γιατί δεν ήταν διαδικτυωμένοι, ε, αλλά όλα αυτά που λέτε μπορούμε να τα δούμε και μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Και αυτά ήταν από δική μου πλευρά. ευχαριστώ. Ο κύριος... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ σύντομο όσον αφορά την ανακαίνιση του Πολ Ανρί Σπακ. Να σας πω ότι όντως οι πληροφορίες που παρέχονται από την Γενική Έκθεση ήταν απλώς μια ενημέρωση για την κατάσταση των πραγμάτων, δεν αποτελούσε έγκαιρη προειδοποίηση, πρώιμη προειδοποίηση τέλος πάντων, αλλά θα έρθουμε με περαιτέρω ενημέρωση και κατόπιν θα έχουμε και αριθμητικά στοιχεία, θα έχουμε πληρέστερα στοιχεία να συζητήσουμε επίσης. Είπαμε για την ε, ανακαίνιση του Στρασβούργου. Επίσης έχουμε το κτίριο, το χώρο της διαπίστευσης και εκεί θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ακούσαμε πολλά, αλλά προτείνουμε επίση να οργανωθούν κάποιες επισκέψεις επιτόπου, ούτω ώστε να είναι ακριβέστερη η εικόνα τη κατάσταση. Πολύ χρήσιμη θα είναι αυτή η επίσκεψη. Uh, Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους τρεις προσκεκλημένους μας. Σίλβα, Περέιρα, Βέλε, Βίλαντ και όσον αφορά το Πολωνρή, ΣΠΑΚ, σίγουρα θέλουμε κάτι να γίνει όσον αφορά περισσότερη ενημέρωση, περισσότερα στοιχεία. Και οπωσδήποτε ενδιαφέρομαστε πολύ για να δούμε τι θα προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.